Uh, well, good afternoon, everybody. Sorry to start the meeting a bit late. I was busy greeting everybody from on return from holiday and I... Σας καλωσορίζω όλους. Για... Μάλλον σας καλωσόριζα όλους έναν ένα και δεν κατάλαβα ότι πέρασε η ώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Βλέπω ορισμένους ιδιαίτερα ηλιοκαμένους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου προέρχομαι τα πράγματα δεν νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ φωτεινά. Πάντως βλέπω ότι δύο μέλη τουλάχιστον ξόδεψαν ένα κομμάτι του χρόνου του στην Ουαλία και στην Αγγλία και αυτό με χαροποιεί. Όχι Άγγλοι βέβαια. Λοιπόν κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτον θα πρέπει να δεχτείτε την ημερησία διάταξη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχέση με αυτό. Στις 3.30 θα έχουμε μια σύντομη ψηφοφορία σε κάποια θέματα, μεταξύ των οποίων και τη νομοδότηση του κυρίου Κοφεράτη. Θα δούμε επίσης και το θέμα το σημαντικό των συμβάσεων παραχώρησης. Η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σας χαιρετώ όλους όσους μας παρακολουθείτε από το δίκτυο. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε δύο νέα μέλη στην Επιτροπή μας. Δεν είναι ακόμα εδώ, αλλά θα τους καλωσορίσω όταν είναι ανάμεσά μας η κυρία Περάρα από τη Γαλλία που αντικαθιστά τον κύριο Αμπάτ και ο κύριος Μάντλενερ ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Στάσεν από την Ολλανδία. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την κυρία Βαντερστάκεν, η οποία είναι νέα υπάλληλος, η οποία ε, γίνεται μέλος της γραμματείας σας καλωσορίζουμε και με χαρά θα συνεργαστούμε. Έχουμε επίσης και τον κύριο Γκρόνμπερ Μέσεν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Δανίας, ειδικό εμπειρογνώμονας ε, στα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν σήμερα. Θα συνεργαστεί και με τον Καλνιόμπολ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε ήδη εμείς εδώ. Ο κ. Γιώργενσεν ήταν και ειδικό σύμβουλος της Προεδρίας της Δανίας. Υπάρχει επίσης ε, έτοιμο ένα σημείωμα ενημερωτικό, το οποίο ονομάζεται για την κατάσταση των πραγμάτων ε, στο θέμα της συνδεσιμότητας ε, του διαδικτύου και της μεταφοράς δεδομένων. Έχει ενδιαφέρον το έγγραφο αυτό, ξόδεψα μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο Silicon Valley στην Καλιφόρνια και έμαθα πολλά για τις εξελίξεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω σήμερα. Θα ήθελα να σας ζητήσω επίσημα να εξετάσετε τα πρακτικά της 20 και 21ης Ιουνίου και θα θεωρηθούν δεκτά τα πρακτικά αυτά μέχρι το τέλος της, της συνεδριάσεως. Το πρώτο κύριο θέμα μας μάλλον σήμερα, βασικό θέμα μας σήμερα, είναι το πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14 με 20. Το λεγόμενο πρόγραμμα Customs, τελωνία. Η κυρία Χάνσλικ θα παρουσιάσει την έκθεση, αν και η συγητής μας είναι ο κύριος Μπαλταζάρη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι το πρόγραμμα αυτό για τα τελωνία μας παρουσιάστηκε σαν ένα μεικτό πρόγραμμα ανάμεσα στα τελωνία και στο πρόγραμμα φυσκάλης για την φορολογία. Υπήρξαν επίπεδα δυσθυμίας υψηλά. Δεν θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο ήταν λογικό. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της για τον συνδυασμό αυτό. Δεν πιστήκαμε και γι' αυτό ζητήσαμε το πρόγραμμα αυτό να γίνει δύο προγράμματα. Ευχαριστώ την Επιτροπή που δέχτηκε λοιπόν την άποψη του Κοινοβουλίου και η κυρία Χάσλιτ θα μας το παρουσιάσει. Έγινε δεκτό από την Επιτροπή στις 29 Αυγούστου και αρχίζουμε την εξέτασή του άμεσα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δώσω το λόγο στην κυρία Χάντσλεκ. Έχουμε τους Χιώδης ε, Μάντελ, Σκοφεράτη και Σμιτ. Και ο ε, Μάντελ είναι εδώ και αυτός. Αλλά όλα τα μέλη που θα ήθελα να ζητήσουν το λόγο μπορούν να το κάνουν. Δίνω το λόγο λοιπόν στη Μαγκρέτα Χάντσλεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόλις ενημερώθηκα από τον κύριο Μπαλτασάρη και γι' αυτό θα σας το παρουσιάσω στα αγγλικά. Στις 29 Φεβρουαρίου του 12 οι συντονιστές της ΣΥΝΚΟ αποφάσισαν να κοπεί στα δύο το πρόγραμμα φυσκάλης της ε, Επιτροπής σε δύο τμήματα, ένα για το τελωνίο και ένα για τα φορολογικά. Συμφώνησαν και οι συντονιστές στις 13 Μαρτίου, ο Επίτροπος Σεμέτα έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ, λέγοντας ότι είναι καλό τα προγράμματα αυτά να παραμείνουν ενωμένα. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή ε, επανήλθε και έλαβε υπόψη της τη θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Στις 29 Αυγούστου λοιπόν η Επιτροπή υιοθέτησε την τροπολογημένη πρόταση για τα τελωνία και για το πρόγραμμα φυσκάλης. Ένα νέο χρονοδιάγραμμα θα παρουσιαστεί στη συνάντηση των συντονιστών της 18 Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις τροπολογημένες προτάσεις της Επιτροπής. Το χρονοδιάγραμμα της αναθεώρησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με την πρόταση για ένα νέο πολιετές οικονομικό πλαίσιο, όπως τροπολογήθηκε στις 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή και με την διαίρεση του προγράμματος σε δύο τμήματα. Δημοσιονομικά μιλάμε για 500 εκατομμύρια, 542 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020, από το 14 μέχρι το 20. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται στην λειτουργία ουσιαστικά της Τελωνιακής Ένωσης. Στόχος των προγραμμάτων αυτών, του προγράμματος αυτού, συγγνώμη, είναι να διευκολύνει την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ολοκλήρωση της Τελωνιακής Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα ακολουθήσει, θα επιδιώξει τις εξής προτεραιότητες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του διοικητικού βάρους και του οικονομικού βάρους και της αντιμετώπισης της τρέβλωσης του ανταγωνισμού της υποστήριξης των τελωνιακών υπηρεσιών στις προσπάθειες τους ε, προστασίας του πολίτη, ε, της ασφάλειάς τους αλλά και του περιβάλλοντος, της βελτίωσης των διοικητικών ικανοτήτων τους και τέλος είναι η καταπολέμηση της απάτης. Αυτό είναι το σημείωμα το οποίο προετοίμασε ο κύριος Μπαλτασάρε και το οποίο σας το παρουσίασα ενημερωτικά. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ας ακούσουμε τα σχόλια των σκιωδών και πρώτος ο κύριος Κοφεράτη. Και εγώ λέω κύριο Σκοφεράτη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τελικά επίστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στον διαχωρισμό. Η προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έλεγα μεθοδολογικά διορθώθηκε και οδηγηθήκαμε σε μια θετική κατάληξη. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια σύντομη βέβαια εξέταση του κειμένου λόγω των προθεσμιών. Υπάρχουν όμως συνθήκες έτσι ώστε να προχωρήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, μιας και η συζήτηση μέχρι τώρα έχει ήδη θα έλεγα ε, υποδείξει τα βασικά προβλήματα τα οποία είναι προς επίλυση. Ε, να πω κάτι τώρα ειδικά για τα τελωνία. Το θέμα των τελωνίων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, σε ένα ευρωπαϊκό γεωγραφικό πεδίο, σαν το ευρωπαϊκό μάλλον, όπου υπάρχει ανάγκη από ένα σύστημα τελωνιακό το οποίο να είναι και αποτελεσματικό και διαφανές στις ενέργειές του και ικανό να παρεμβαίνει με ταχύτητα. Ο έλεγχος ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο αυτοματισμένα και εδώ απαιτείται και αύξηση των πόρων όπως ακριβώς προτείνεται είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τους πολίτες να επιλέξουν με σωστό τρόπο τις, να κάνουν τις επιλογές στον εθνικό χώρο τον οποίο έχουν ακριβώς στον οποίο εθνικό χώρο βρίσκονται. Πρέπει λοιπόν μέχρι το 2020 να πιέσουμε έτσι ώστε οι διαδικασίες να αυτοματοποιηθούν ακόμα περισσότερο και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε με συστηματικό και συνεχή τρόπο τις διαδικασίες ελέγχου. Ένα άλλο θα έλεγα ειδικό θέμα το οποίο θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε σε άλλη φάση είναι η αντιμετώπιση των απατών και των απατών στις εμπορικές συναλλαγές και των απατών σχετικά με την λεγόμενη πολιτιστική παραγωγή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε και να αξιολογήσουμε σωστά τα θέματα που άπτονται των συγγενικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είμαστε σωστότερα ενημερωμένοι για να αποφύγουμε τα λάθη τα οποία θα μπορούσαν να, να μας οδηγήσουν σε παλινοδίες αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Σε αυτή τη φάση απλά ήθελα να υπογραμμίσω τη χρησιμότητα και το έφθετο του διαχωρισμού και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ειδικά για τα τελωνία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Μάντερς, στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εύχομαι και εγώ το... Καλώς ορίσατε σε όλες και όλους. Ο συνάδελφός μου με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω. Ήθελε να βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, α, είναι αριθμός δημοκράτης ή δημοκρατικό, δεν δημοκρατικό, αποφάσισα λοιπόν η Κομισιόν να χωρίσει τα προγράμματα σε φυσκάλης και τελωνίων, όπως είπαν οι άλλοι προηγούμενοι συνάδελφοι, γιατί αυτό θα προκαλέσει λιγότερη σύγχυση στις ε, δικαστικές αρμοδιότητες. Πάνω όλα αυτά, ε, μας αρέσει η πρόταση. Θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμη για τις χώρες μέλη. Για τα τελωνία χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Άλλωστε είναι και πιο δίκαιο το σύστημα αυτό για τα εξωτερικά σύνορα. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένε ανησυχίε. Η Κομισιόν προτείνει φιλόδοξη πολιτική επιλογή για το τμήμα των τελωνίων. Ο κ. Σμιτ ο συνάδελφος δικαστητό, θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκή κονδύλια, νέα συστήματα μηχανογράφησης και εξυγχρονισμό των τελωνίων. Οι χώρες μέλη μάλλον δεν θα συμφωνήσουν, διότι βέβαια θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τους αρέσει, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Η Κομισιόν πρέπει να φροντίσει ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις πιο χρήσιμες επιλογές. Ο δεν θεωρεί ότι, δεν είναι πεπισμένος ότι χρειάζεται ειδικό οργανισμός για τα τελωνία, διότι ενδέχεται να επικαλυφθεί το έργο της με το έργο άλλων υφισταμένων οργανισμών. Και αυτό βέβαια θα πολλαπλασιάσει τα έξοδα. Αυτά ήθελε να πει ο Όλε Σμιτ και ευχαριστεί όλες και όλου που συνεργάστηκαν μαζί του. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί, ρωτά ο πρόεδρος. Καλωσορίζω και την ομάδα της Επιτροπής, ο κύριος Δασκάλου. Είναι παρόν, ο κύριος Ντεγράφ. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Εσείς. Ο κύριος Δασκάλου, αν δεν κάνω λάθος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για την υποστήριξη που προσφέρετε στο νέο πρόγραμμα και που το βάλατε και τόσο σύντομα στην ημερήσια διάταξή σας. Το νέο πρόγραμμα Τελωνίων 2020 και πώς συγκρίνεται με αυτό που ισχύει μέχρι τώρα. Σχεδιάσαμε το νέο πρόγραμμα βασισμένοι στα στοιχεία που απέδωσαν μέχρι τώρα και που αποτελούν την αξία του τρέχοντος προγράμματος, τα πήραμε υπόψη αυτά, ώστε το νέο νομικό κείμενο να περιλάβει τα βασικά στοιχεία του υφιστάμενου προγράμματος και να τα επεκτείνει όπου αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσει σωστά τις ε, προσδοκίες από τώρα μέχρι το 2020. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ ανοιχτοί και ιδίω σε ό,τι αφορά τους εποφελούμενους το πρόγραμμα του 2020 καλύπτει τους νυν δικαιούχους, δηλαδή κυρίως τις χώρες μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες της πολιτικής γειτονίας. Αυτές οι χώρες μπορούν να συμμετέχουν βέβαια κατά περίπτωση, αλλά όχι σε όλο το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους, ίσως υπάρχει μια διαφορά με αυτούς του προγράμματος φίσκους, αλλά όταν τα εξηγήσαμε αυτά, ίσως ήταν μια διαφορά στην παρουσίαση, γιατί οι στόχοι είναι ακριβώς ίδιοι. Για τεχνικούς λόγους και για να ευθυγραμμιστεί η ορολογία με όλα τα προγράμματα της Επιτροπής, βάλαμε ένα σετ ενός με στόχου, κάποιων γενικών στόχων και κάποιες προτεραιότητε. Αλλά σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο είναι ακριβώς ίδιο. Υπάρχουν νέα στοιχεία στις επιλέξιμε δράσεις με τρεις κατηγορίες μία που είναι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, που είναι και το σύστημα μηχανογράφητης, είναι, αυτό το λέμε IT Capacity Building, γιατί είναι πολύ πιο φιλόδοξο από το πρόγραμμα που είχαμε πριν και θα σας πω γιατί. Δεύτερη κατηγορία είναι οι κοινέ δράσεις για την δημιουργία ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τέλος ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση των αξιωματούχων. Υπάρχει και ένα νέο εργαλείο το οποίο εισαγάγαμε στη νέα πρόταση. Είναι η τεχνογνωσία, δηλαδή η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που οφείλεται, βασίζεται μάλλον, στην επιθυμία πολλών χωρών μελών να συμβάλλουν όλες οι χώρες με την τεχνογνωσία που διαθέτουν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ταχύτερα και φθηνότερα ένα ενίο σύστημα. Με κοινέ δηλαδή προδιαγραφές, να δημιουργηθούν δηλαδή κοινέ προδιαγραφές ή να συμβληθούν οι διάφορε τεχνογνωσίες για να αντιμετωπιστούν οι διάφορε επιχειρησιακές ανάγκες. και ειδικέ δραστηριότητες για ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. Το ίδιο και για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. Εμπνεώμαθα λίγο από το πρόγραμμα Φισκάλης, από τα φορολογικά. Ορισμένε χώρες χρειάζονται κάποια διοικητική υποστήριξη και από το πρόγραμμα του 2013, μέχρι το 2013 δηλαδή, όπου έχουν συμπεθεί ορισμένα προβλήματα. Το εργαλείο αυτό φαίνεται να είναι επιτυχές στο πρόγραμμα Φισκάλης. Επειδή τώρα κινούμεθα προς την κατεύθυνση του μελλοντικού σχεδιασμού των επόμενων 7-8 χρόνων, είναι σκόπιμο να μπουν αυτές οι δραστηριότητες στην πρότασή μας. Καταργήσαμε επίσης ε, τις ε, δράσεις benchmarking, όχι επειδή δεν χρειάζονται, αλλά διότι θεωρήσαμε ότι με το εργαλείο που διαθέτουμε μπορούμε να καλύψουμε σιωπηρά το benchmarking και τη steering group που είναι μονάχα ενός είδους steering groups. Αυτά σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δράσεις, αυτές είναι οι βασικές αλλαγές. Θα δείτε ότι σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό δεν έχει αλλάξει αυτό που ζητούμε σε σχέση με το τμήμα το φορολογικό του προγράμματος φίσκους. Ακολουθείτε η διαδικασία εξετάσεως και θα χρησιμοποιηθούν και ετήσια προγράμματα που θα εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή σε ετήσια βάση. Είναι πιο εξελιγμένο το πρόγραμμα σε σχέση με το τρέχον μέχρι το 2013 και όλοι αναμένουμε ότι θα είναι και πιο έντονο το στοιχείο της απόδοσης λογαριασμού. Αυτά είναι οι βασικές γραμμές του νέου προγράμματος. Με λίγα λόγια, το νέο πρόγραμμα ακολουθεί γενικά τις γραμμές του τρέχοντος προγράμματος χωρίς μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν προβλέψεις για κάποιες νέες δραστηριότητες σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε για τη μελλοντική εξέλιξη του τελωνιακού έργου στο, στις ευρωπαϊκές κοινότητες για το μέλλον και αυτά. Ευχαριστώ για την χρήσιμη σύνοψη λέει ο Πρόεδρος, ως γνωρίζετε η παρούσα Επιτροπή υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας πολύ αποτελεσματικής τελωνιακής υπηρεσίας και όπως έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι. Και ο κ. Μπαλτασάρε είμαι βέβαιος ότι θα εξετάσει προσεκτικά στη συνεργασία με τους και συγιτές το θέμα αυτό και για την επόμενη εξέταση του θέματος. Ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα που έχουμε μπροστά μας, έχουμε χρονοδιάγραμμα. Όχι. Καλά. Οι συντονιστές θα επανεξετάσουν το χρονοδιάγραμμα σε λίγες εβδομάδες, αλλά θα κινηθούμε όσο γίνεται ταχύτερα με την συνεργασία του κ. Μπαλτασάρε. Επιθυμεί κανείς να συμπληρώσει ή να ε, παρατηρήσει κάτι. Όχι, σας ευχαριστώ λοιπόν. Καλά. Και τώρα προχωρούμε, είμαστε ακριβώς στις 3.30, στις ψηφοφορίες του σημερινού απογεύματος. Άρα, πρώτα έκθεση De Jong, μετά Κοφεράτη και μετά Ροσφόρ. Αυτέ, ορισμένες από αυτές έχουν σχέση με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων τριμερού διαλόγου. Πρώτα λοιπόν θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση De Jong, τμήμα τρίτο, για το προπολογισμό του 2013. Θα δώσω το λόγο στον κύριο De Jong για να κάνει την εισαγωγή στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα παρέμβω σύντομα. Είχαμε καλή συνεργασία για τον προπολογισμό. Έλαβα διάφορες προτάσεις για τροποποίηση των ίδιων των γραμμών του προπολογισμού και μπορέσαμε να φτάσουμε σε συμφωνία για διάφορες συμβιβαστικέ. Υπάρχει προφορική τροπολογία για μία συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού Νομίζω όμως ότι πρώτα θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση και οπότε θα τα αφήσω αυτό το σχόλιο για αργότερα. Μάλιστα. Θέλετε να μιλήσετε τώρα για τη γραμμή του προπολογισμού ή μετά σας δώσω το λόγο στην γνωμοδότηση, όπως θέλετε εσείς. Ωραία. Ας κάνουμε τότε πρώτα την γνωμοδότηση. Είναι όλοι ικανοποιημένοι και έτοιμοι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε κάρτες ψηφοφορίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν τις έχετε, καλό είναι. Πάντως, σας βλέπω τους ή άλλους, διαφορετικά θα μετρήσουμε. Για τον κατάλογο ψηφοφορίας, λοιπόν, έχουμε την συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σαφώς. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 12 του κυρίου Χαμών. 12 υπέρ. Υπέρ, ας μετρήσουμε. Πάνω τα υψηλά τα χέρια, όσοι ε, είστε υπέρ. 8. Κατά. Κατά. 12. Αποχές. 3. 4. Ωραία. Απορρίπτεται. Στο φίτσι, Uh, Amendment 13, Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. De Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πέντε de Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 14. Η 12 δεν εγκρίθηκε, άρα ψηφίζουμε για την 12. 14. Ποιοι είναι υπέρ, ή κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε λοιπόν τις γραμμές του προπολογισμού, πρέπει να τις συζητήσουμε. Θέλεις να πεις κάτι? Ναι, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το κείμενο είναι σωστό όπως έχει υποβληθεί. Απλώς θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι για το Solvit ζητάμε 1,3 εκατομμύρια. Γιατί σε προηγούμενες εκδοχές έγραφε ένα επιπλέον εκατομμύριο σε σχέση με τη τωρινή γραμμή. Όπω το έχω εγώ τώρα και το έχει μπροστά η Επιτροπή είναι σωστό και αντιπροσωπεύει τα τελευταία διαπραγμάτευση. So if we, if we go through this um, Ωραία λοιπόν να ψηφίσουμε κάθε σειρά χωριστά. Yeah. So I'll, Θα σας λέω το νούμερο της γραμμής κάθε φορά. Λοιπόν, Γραμμή 6900. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εκτός θα μετράω την κυρία Χάνσλι, κάποιος άλλος που δεν έχει την κάρτα. Γιατί έχουμε αρκετά να κάνουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 6900.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 Vote. Anyone who not voted? No. The vote's closed. The vote is closed. So that's 18. Τέλος ψηφοφορίας. 18 κατά. Απορρίπτεται. 6.903. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 ψήφι υπέρ και 13 κατά. Τροπολογία 6904 με προφορική τροπολογία που νομίζω το έχετε κάτω-κάτω στον κατάλογο ψηφοφορίας. Την έχετε αυτή την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτει 6.905 και πάμε στην 6.907 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε την 6.906 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έτσι. Τελειώσαμε τις γραμμές του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ, Ντένις. Ντε Θέλεις να πεις κάτι ακόμα? για το επόμενο βήμα στη συζήτηση περί προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ε, έχει προβλεφθεί συνεδρίαση για τις 18 Σεπτεμβρίου όπου θα συνεδριάσουμε όλοι οι συγκητές των διαφόρων επιτροπών και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να υπερασπιστούμε φυσικά τις τροπολογίες που μόλις εγκρίναμε. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ λοιπόν ώστε να περάσουν όλες αυτές οι τροπολογίες. Μάλιστα, ωραία. Ναι, ξέρουμε ότι θα υποστηρίξει την θέση μας για τον προπολογισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και προχωράμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Κοφεράτη προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Αγορά για τις ε, κάρτες στο ίντερνετ και τις κινητές, πληρωμές μάλλον από κινητά τηλέφωνα. Ο κύριος Κοφεράτη, επειδή αν θέλουν κάποιοι σχεδόν να παρέμβουν και μετά θα περάσουμε σε ψηφοφορία. Εγώ θέλω μόνο να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους συνεργαστήκαμε καλά. Νομίζω πως τα βασικά προβλήματα λύθηκαν μέσω των συμβιβαστικών ε, τροπολογιών. Παραμένουν κάποιες αποκλήσεις απόψεων για ένα-δυο πτυχές, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν πως το σύνολο του νομοδότηση θα μπορέσει να εγκριθεί και αντιστοιχεί στους προσανατολισμούς που συζητήσαμε στη διάρκεια των περασμένων μηνών. Εγώ είμαι ικανοποιημένο από την ε, διαθεσιμότητα και από την προσοχή που, έδωσαν, που έδειξαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει? Right. Let's move on to the vote, then. Ας περάσουμε στη ψηφοφορία. Όλοι είναι εξοπλισμένοι με κάρτες, οπότε αν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε, εκτός από την κυρία Χάνσλικ. 1 του εισηγητή υπέρ, κατά εγκρίνεται. 2 προσθήκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. 3 αρίας υπέρ, κατά εγκρίνεται. 4 αρίας υπέρ, κατά εγκρίνεται. 5 τουν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. The vote closed and that's carried. Εγκρίνεται 18 προς 11. 6 Άριας, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 το εισηγητή, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 Άριας, Σβάμπ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Άριας, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12 το εισηγητή, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 19 τουν υπέρ κατά εγκρίνεται 20 έχει αποσυρθεί συμβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην τροπολογία 28 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται 30 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 29 Σαλβίνη υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική νομίζω πως όλες καταπίπτουν ναι ε, τροπολογία 34 έγκστρομ υπέρ κατά εγκρίνεται 35 υπέρ Τροπολογία 35, Έγκστρομ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη ψηφοφορία της τροποποιημένης ε, γνωμοδότησης, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν για το σύνολο της γνωμοδότησης. Τέλος της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, 2 κατά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοφεράτη. Και Φυσικά θα υπερασπιστείτε τις απόψεις μας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Και τώρα περνάμε για την εντολή, να συζητήσουμε μάλλον για την εντολή για τις ε, διαπραγματεύσεις. Θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει με τους συζητητές. Ε, καταρχήν ε, είχαν έρθει να το συζητήσουμε στους συντονιστές και μετά αποφασίσαμε ότι έπρεπε να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή. η Επιτροπή πρέπει αυτό να το εγκρίνει. Χρειαζόμαστε 21 ψήφους δηλαδή υπέρ της εντολής. Αν κανείς σκεφτόταν να φύγει, να σας πω δηλαδή ότι χρειαζόμαστε την ψήφο σας. Θα ζητήσω από τον κύριο Ρόσφορντ να μας παρουσιάσει, να συνοψίσει τη θέση του. Νομίζω πως είναι καλό αυτό γιατί θέλουμε όλα αυτά να έχουν καταγραφούν. Ο κύριος Ρόσφορντ λοιπόν και αν κανείς άλλος θέλει να σχολιάσει μπορεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια μόνο. Η έκθεση αυτή, η οποία αφορά τους καταναλωτές, τη συζήτησαν οι συντονιστές τον μήνα Ιούλιο. Ενέκριναν την ιδέα του να ξεκινήσουμε ανεπίσημες διαπραγματεύσεις και επί τη βάση αυτής της συνεδρίασης των συντονιστών θα καθοριστεί το αντικείμενο της εντολής διαπραγμάτευσης. Δεν θα μπούμε σε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι όπως και οι συντονιστές και όσοι στην Επιτροπή εγκρίνουν τη διαδικασία αυτή, εφόσον το επισημοποιήσουμε θα ξεκινήσουμε τεχνικές συναντήσεις τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω εδώ. Καλώς. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική μέθοδο. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε απλά ξεχάστε το ποιος είναι υπέρ. Ψηφίζετε. Καλώς πέρα της ψηφοφορίας. «24 υπέρ, μία αποχή, έχετε την εντολή διαπραγμάτευσης πλέον». Οι συγητή και οι σκιώδεις συγητέ είναι η ανεπίσημη διαπραγματευτική ομάδα και εγώ και οι αντιπρόεδροι θα προεδρεύσουμε των διαπραγματεύσεων. Το επόμενο θέμα έχουμε ξεχωριστές ψηφοφορίε για τα δύο επόμενα θέματα. Θα δώσω το λόγο στον Γκρέκ πρώτα. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει μετά για την εισηγήτρια του ΕΛΚΑ. Ίσως ο κύριος Γκρέκ βέβαια να μπορέσει να μας μιλήσει και για τις δύο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην έγκριση σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δεχτούμε άμεσα τα πάντα. Εμείς πιστεύουμε ότι η επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς είναι κάτι το καθοριστικό για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου λοιπόν Θέλουμε η απόφαση να ληφθεί ταχύτατα. Πρέπει να πούμε ότι εάν διαπιστώνουμε ότι οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν γίνονται σεβαστές και δεν διαφυλάσσονται, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Αυτή πρέπει να είναι η θέση μας. Καλώς. Μία σύντομη έκθεση. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Τι πιστεύει. Εγώ το υποστηρίζω κατά βάση, αλλά με ενδιαφέρει εάν το Συμβούλιο ήδη έχει εγκύψει. Ο κ. Γκρέσ. Οι, οι επίσημες πληροφορίες που έχω μάλλον ανεπίσημες πληροφορίες που έχω μου λένε τι πιστεύει το Συμβούλιο αλλά η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει αργότερα. Όταν θα την έχουμε αυτήν θα συζητήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και βέβαια πού βρίσκονται τα απολύτως ανυπέρβλητα όρια μας. Ο Πρόεδρος. Το Συμβούλιο πρόσφερε τη δυνατότητα να ε, ε, εισέλθουμε σε διαπραγματεύσεις και αυτό θα συζητήσουμε και με τους συντονιστές. Ας, ας ψηφίσουμε από κοινού λοιπόν και για το ADR και το ODR. Resolution for a mandate. Um, the vote is open on the a mandate for uh, the Mr. report. Λοιπόν, η έκθεση του κυρίου Γκρέκ πρώτα. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ. Κύριε Γκρέκ, έχετε την εντολή που θέλατε. Η δεύτερη έκθεση για τις ρυθμίσεις online. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ μία εποχή. Λοιπόν, θα οργανώσουμε τους τριμερούς διαλόγους, τριμερείς, συγγνώμη, διαλόγους. Θα αποφασίσει η διαπραγματευτική ομάδα το πώς θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι καλό θα είναι όλοι οι συγητές να είναι παρόντες στη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων. θα προεδρεύω ή εγώ όπως είπα ή ένας από τους αντιπρόεδρους μας. Καλώς. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε είναι τα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για μια όχι ιδιαίτερα συνηθισμένη διαδικασία λόγω του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είναι η αρμόδια επιτροπή. Δεν ξέρω, έχουμε υιοθετήσει τις τροπολογίες, διαρωτάται ο Πρόεδρος. Έχουν προετοιμαστεί οι τροπολογίες από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Θα ψηφίσουμε στις 18 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, η ευκαιρία την οποία έχουμε τώρα είναι να ακούσουμε τα σχόλια τα οποία θα ήθελα να κάνουν οι συνάδελφοι για τις τροπολογίες. Και ίσως στην αρχή να ζητήσω από αυτούς που έχουν καταθέσει και συντάξει τις τροπολογίες να μας πούν τη γνώμη τους. Ο κύριος Γκρέκ. Αν χρειαστεί θα ακούσουμε και σχόλια από συναδέλφους. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για να προετοιμάσουμε σωστά ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και γι' αυτό εμείς καταθέσαμε τις τροπολογίες αυτές. Θεωρώ ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να ακολουθεί ένα από τα βασικά, θα πρέπει να παραμείνει ένα από τα βασικά κριτήρια των στόχων για το 2020. Η ενιαία αγορά είναι βασικό μέσο για να ξεπεράσουμε την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Έτσι θα δημιουργήσουμε περαιτέρω ευημερία και κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ κύριε Γκρέκ. Καλό είναι που επιστήσατε την προσοχή μας στις εκθέσεις μας τις παλαιότερες, ιδιαίτερα αυτήν στην οποία αναφέρατε την ενιαία αγορά. Κύριε Ρούλε, θέλετε το λόγο. Όχι. Κύριος Μάντερς έχει καταθέσει το απολογία. Θέλετε να μιλήσετε κύριε Μάντερς. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να επικοινωνεί καλύτερα το τι σημαίνει η εσωτερική αγορά. Είναι το θεμέλιο η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενημέρωση προς τους πολίτες πρέπει να είναι σωστή. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφημίσει την εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι η κατέθεσαν ανθρωπολογίας δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο πριν ψηφίσουμε, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία την επόμενη φορά. Να πω ότι το θέμα το συζητήσαμε σε επίπεδο συντονιστών και θα το συζητήσουμε και στο τέλος Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε δηλαδή τη μελλοντική, για τη μελλοντική δομή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το πώς στην εσωτερική αγορά θα ενταχθούν καλύτερα τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Εδώ τίθενται θέματα συντονισμού περισσότερο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, θα έλεγα, πιστεί για την προώθηση της εσωτερικής αγοράς και τον ρόλο των καταναλωτών. Νομίζω ότι η ιδιαίτερη έκθεση του κυρίου Γκρέκ απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξουν συγκεκριμένες αναφορές σε κάποια από τα έγγραφα τα οποία έχουμε ήδη εξετάσει θα τα δούμε αυτά καλύτερα και σε επίπεδο προέδρων πολιτικών ομάδων για να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στα πλαίσια του επομένου κύκλου, το 2013, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για την εξέταση του θέματος αυτού. Αποκινούμε τους συντονιστές έτσι ώστε να κάνουμε και τις κατάλληλες προτάσεις. Καλώς λοιπόν κλείνουμε το θέμα αυτό τώρα. Έχουμε πάει σχετικά γρήγορα και μιας και ο κύριος Κοφεράτη είναι εδώ. Θα ήθελα να ελέγξω αν έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι βέβαια. Να διακόψουμε για μισή ώρα λέει ο πρόεδρος. Δεν θα έρθει πριν τις 5 λοιπόν και η Επιτροπή δεν είναι εδώ. Θα διακόψουμε για μισή ώρα. Ζητώ συγγνώμη που καθυστερώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς στις και μισή με την έκθεση Κοφεράτη.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

All right, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for, for waiting and for Mr. Kofferati's patience. Ευχαριστώ τον κύριο Κοφερέτη για την υπομονή του. Ο κύριος Σαρτρέν είναι εδώ. Όχι, ο κύριος Ρόιτερς τελικά, ο οποίος είναι τμήματάρχης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ήταν και στην Επιτροπή Μεταφορών πριν από εδώ, έχει πολλή δουλειά. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στη γνωμοδότηση Κοφεράτη, στα πλαίσια των δικτύων. Έχουμε μαζί μας τον εισήγητη, η κυρία Χάνσλεκ θα πάρει το λόγο για το ΕΛΚ. Εργάζεται πολύ σκληρά η κυρία Χάσλετ. Δεν ξέρω κάποιος άλλος από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, όχι. Λοιπόν, τότε θα έχουμε μια γενική συζήτηση. Ο εισηγητής λοιπόν θα σχολιάσει τις τροπολογίες τις οποίες έχει λάβει και μετά θα ακούσουμε από τους ε, εισηγητές θα ζητήσουμε και από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να κάνει τα σχόλιά του και μετά θα επανέλθουμε στον κύριο Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο τοπολογίες εδώ. Molto tempo per commentarli perché una parte consistente di questi emendamenti 72 si υπάρχουν ένα τμήμα των τροπολογιών αυτών ε, ε, Λοιπόν, είναι τροπολογίες οι οποίες γενικά είναι θετικές στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο την ενίσχυση, την κατεύθυνση η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία σχολιάσαμε στις προηγούμενες συζητήσεις. Κάποιες από τις τροπολογίες αυτές περιλαμβάνουν ορισμένες διατυπώσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα θα έλεγα ξεκάθαρες και κατανοητές. Εγώ θα προσπαθήσω να κατανοήσω τις πραγματικές προθέσεις αυτών που καταθέτουν τις τροπολογίες. Θα το κάνω αυτό σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές ή και άμεσα με αυτούς που καταθέτουν την τροπολογία, αμέσως μετά αυτήν εδώ τη συζήτηση. Θα ήθελα με τη σημερινή συζήτηση να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλα προβλήματα, τα οποία έστω και με διαφορετικό τρόπο έχουν γίνει αντικείμενο τροπολόγησης. Πρόκειται για δύο σημαντικά θέματα, τα οποία απαιτούν την προσοχή μας. Τα εξής. Το πρώτο αφορά την ευελιξία στη χρήση των όρων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει δύο προθεσμίες. Το 2030 για το κεντρικό δίκτυο, το λεγόμενο Core Business, και το 2050 για το σφαιρικό δίκτυο. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν θεωρήσει ότι οι ενδείξεις αυτές είναι υπερβολικά άκαμπτες και ως εκ τούτου θεωρούν ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν. Θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά βέβαια συγκεκριμένα με αυτούς που κατέθεσαν τις τροπολογίες. Πάντως πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχει κανείς χρονικές αναφορές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις πιθανές δυσκολίες οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν στην πορεία σε κάποια χώρα στην προσπάθεια σεβασμού των προθεσμιών που θέτει η Επιτροπή, η Οδηγία. Πιστεύω λοιπόν ότι η συμβιβαστική προσπάθεια την οποία εμείς θα πρέπει να κάνουμε θα είναι η εξή και σε επίπεδο ενιολογικό αλλά και γενικότερο. Θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε επί της ουσίας τις προθεσμίες και ταυτόχρονα να προβλέψουμε τις περιπτώσεις και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη χορήγηση παρεκκλήσεων ή εξαιρέσεων θα πρέπει δηλαδή εμείς να καταστήσουμε το μη σεβασμό των προθεσμιών εξαίρεση και όχι να καταστήσουμε ικανές τις χώρες συνειδητά να προσπαθήσουν να λειτουργούν χωρίς χρονικές προθεσμίες. Γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο αυτό δεν θα γνωρίζουμε ακριβώς ε, ε, πώς είναι η κατάσταση ιδιαίτερα για τις νέες χώρες αλλά μία κάποια λοιπόν ευελιξία είναι σωστό να υπάρξει σαν ε, ιδέα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει κανόνας. Το δεύτερο μεγάλο πλαίσιο είναι το λεγόμενο governance, διακυβέρνηση στην διαχείριση των διαδρόμων. Όπως είπαμε την τελευταία φορά, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο των συντονιστών. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα ποιες είναι οι αρμοδιότητες των συντονιστών και οι τρόποι συντονισμού των αρμοδιοτήτων αυτών. Αυτό έτσι ώστε οι συντονιστές να έχουν μια ουσιαστική, να χαίρουν μια ουσιαστική αυτονομίας, αλλά να μην επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες τους, όπως βλέπω εγώ τουλάχιστον και το εννοώ έτσι διαβάζοντας τις τροπολογίες τους, να μην αντικαθιστούν οι συντονιστές τις κρατικές αρχές. Είναι όμως προφανές ότι όταν πρέπει κανείς να δημιουργήσει κάποια έργα, υποδομές με αρκετά μεγάλη σημασία που καλύπτουν ή συνδέουν αρκετά μεγάλα εδάφη, είναι σίγουρα απαραίτητο να υπάρξει μία υπερεθνική αρχή έτσι ώστε να μπορεί να επιλύει τις αντιφάσεις που δημιουργούνται, τις διαφορές που δημιουργούνται ή να ξεπεράσει τις δυσκολίες τις οποίες θα συναντά κανείς ε, στην πορεία. Γι' αυτό λοιπόν η πιθανή λύση σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι η εξής όχι να αφαιρέσουμε αρμοδιότητες μεν από τους συντονιστές, αλλά να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, έτσι ώστε να μην αντιτίθενται και να μην επικαλύπτονται με τις αρμοδιότητες των τοπικών και εθνικών αρχών. Νομίζω ότι δεν θα συνεχίσω. Νομίζω ότι παρουσίασα ποια είναι τα δύο βασικά θέματα, τα δύο βασικά προβλήματα. Αυτά θα πρέπει να αναζητήσουμε, να καλύψουμε με συμβιβαστικές προτάσεις. Τα υπόλοιπα είναι εύκολο να ξεπεράσουμε. Good. Okay. Well, thank you very much indeed. Um... Ευχαριστώ πολύ. κυρία Χάνσλικ. Έχετε καταθέσει πολλές τροπολογίες. Σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα δηλαδή. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ τη κυρία Ηλιάνα Ιβανόβα, θα ήθελα να σε χαρώ τον εισηγητή κύριο Κοφεράτη για το εξαίρετο έργο του. Όλοι έχουμε κοινό στόχο να ανταποκριθούμε περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών και να διευκολύνουμε την ομολή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε για τα συγκεκριμένα βήματα ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να πλαισιώσουμε τους στόχους μας. Η κυρία Ιβάνοβα υποστηρίζει την έκθεση του κυρίου Κοφεράτη στη γενική της προσέγγιση και ιδιαίτερα όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους χρήστες, τη βελτιωμένη και τη βελτίωση και την προώθηση της ασφάλειας των δρόμων. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόταση, η κυρία Ιβανόβα πιστεύει πως θα ήταν πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για διάφορα θέματα τα οποία προτείνει η ομάδα του ΕΛΚ. Έτσι θα αποφύγουμε τη δημιουργία επιπλέον ε, διοικητικού φόρτου για τα κράτη-μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται, καθώς και μη ε, απαραίτητες και δαπανηρές ε, διαδικασίες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τονίζουμε την ε, δυνατότητα πρόσβασης στις ε, αεροκατοικημένες περιοχές. Οι πολίτες μας θα πρέπει να είναι ε, σε θέση να χαίρουν τις ελεύθερες κυκλοφορίες ανεξάρτητα από το πού κατοικούν γεωγραφικά. Τρίτον, η δημιουργία μιας κοινή ε, ευρωπαϊκής πλατφόρμας μεταφορών θα πρέπει να συμβαδίζει με αυτόν τον κανονισμό έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διατάξεις από την άποψη των χρηστών. Θα πρέπει να προσφέρονται στους ε, επιβάτες ε, προσβάσιμες πληροφορίες με τυποποιημένη διαδικασία έκδοσης και τιμολόγησης των εισιτηρίων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα εισιτήριο για διασυνοριακά διασυνοριακές μετακινήσεις, εισιτήριο που θα ισχύει για διάφορα μέσα μεταφορών. Αυτή η πλατφόρμα θα λαμβάνει και τα παράπονα των χρηστών και θα πρέπει να εμπνέεται από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές στα κράτη-μέλη στον τομέα των μεταφορών. Πρόκειται για μια πρακτική που θα έχει προστιθέμενη αξία για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Σε σχέση με τις ε, προθεσμίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2013 30 μάλλον για την ολοκλήρωση του βασικού πλαισίου και μέχρι το 2050 για την ολοκλήρωση του πλήρους δικτύου. Ωστόσο, δεδομένης της κρίσης που σοβεί σε διάφορες χώρες, θα πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική ώστε να συμπεριλάβουμε κάποιες εξαιρέσεις στις διατάξεις του κανονισμού μας ή να καταστήσουμε την ε, προθεσμία πιο ευέλικτη. Η κυρία Ιβανόβα θεωρεί ότι τα βασικά σημεία του ΕΛΚΑ θα γίνουν δεκτά και θα μπορέσουμε να έχουμε μία κοινή κατανόηση για τα θέματα που μπορεί καταρχήν να φαίνονται αντιφατικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή είναι η άποψη της κυρίας Ιβανόβα, που είναι η σκαιόδηση Uh, Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χάνσλικ. Κύριε Μάντε, και ξέρω και ότι η κυρία Ρούλη είναι σκιώδη. Κύριε Μάντε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Oh, Ή να δώσω πρώτο λόγο στην κυρία Ρούλε που είναι σκιώδη για το θέμα για του πράσινου. Ευχαριστώ και υποστηρίζω τον εισηγητή στην ιδέα που έχει να αναθέσει στους συντονιστές την διοργάνωση του διαλόγου. Και απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να σκεφτεί ότι τα μεγάλα έργα μεταφορών έχουν συζητηθεί όλο και περισσότερο. Εάν τελικά ο σχεδιασμός δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω του ότι δεν υπάρχει επαρκής διάλογος, αυτό απλώς κοστίζει παραπάνω. Γι' αυτό θα ήμουν ιδιαίτερα γνώμων εάν επανεξετάσουν την θέση τους. Έχω το παράδειγμα της Στουτγάρδης. Εάν είχε γίνει εγκαίρος ο διάλογος με τα θυγόμενα στρώματα του πληθυσμού, θα είχαν αποφευθεί πολλές συγκρούσεις. Όταν όμως αφήνουν και περνά καιρός και γίνονται ζυμώσεις, τα πράγματα δυσχεραίνονται όλο και περισσότερο. Ίσως λοιπόν ένας διάλογος να φανεί εκ πρώτης όψεως ότι προκαλεί κάποια δυσχέρεια, μετά όμως μακροπρόθεσμα αποδίδει. Μάντερς, θέλετε να πείτε τίποτα? Για, πάλι για το για λογαριασμό του κ. Σμιτ. Ναι. Είναι σημαντικό θέμα. Και από ό,τι λένε οι συνάδελφοί μου εδώ, είναι σημαντικό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχω και εγώ μια ενημέρωση από τον κύριο Σμιτ που λέει ότι θα σα το διαβάσω. Συμφωνεί με τον εισηγητή σχετικά με τον ρόλο των συντονιστών. Είναι σημαντικός ο, ο ρόλος του συντονιστή για, τον, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Συμφωνεί με τα όσα έχει πει για τις ε, βιώσιμες μεταφορές. Θεωρεί όμως ο κ. Σμίτ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα και να ενισχυθεί η τεχνολογική καινοτομία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα και στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην, ε, στα σημεία εχμής. Δεν μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε την οικονομική κατάσταση που θα ισχύει στο 2030 ή 2050, αλλά πρέπει πάντως τώρα να κινητοποιηθούν οι χώρες μέλη και να ε, καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Και ο κύριος Σμιτ ευχαριστεί όλους και όλους για τη συνεργασία τους. Uh, uh, Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ. Άλλος κανείς, άλλος ή άλλη βουλευτής. Μήπως τότε η Κομισιόν. Λίγα για την πρόταση, κύριε Ρόιτερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αντιδράσει στη συζήτηση. Πράγματι έρχομαι από την Επιτροπή Τραν, όπου συζητήσαμε το θέμα αυτό και τέθηκε το θέμα ιδιαίτερα των διαδρόμων. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Επιτροπής για την έκθεση Κοφεράτη, όπως σας είπε και ο κ. Σαντράν σε μια προηγούμενη συνάντηση, είναι μια εξαιρετική έκθεση η οποία υπογραμμίζει με σωστό τρόπο τα θετικά της προτάσεως της Επιτροπής. Βλέπουμε ποιες είναι οι αντιδράσεις στις τροπολογίες των διαφόρων μελών και καλωσορίζουμε τις περαιτέρω προτάσεις, ιδιαίτερα στην εδαφική κατανομή, στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες στις οποίες θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί και να μην προχωρήσουμε σε αντιφάσεις με αυτά που λέει η έκθεση. Όπως είπε και η κυρία Χάνσλε και ο κύριος Μάντελ, θα πρέπει να είναι ισχυρός ο ρόλος των συντονιστών. Είναι κάτι το πολύ θετικό, απεδείχθη τον τελευταίο καιρό σαν κάτι το ιδιαίτερα επιτυχές. Αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Παράλληλα, οι προθεσμίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές χωρίς προθεσμίες δεν θα υπάρξει δίκτυο. Εργαζόμεστε προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία 20 χρόνια και βλέπουμε ότι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν τηρούνται. Στο άρθρο 50 θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε μια κάποια ευελιξία την οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεώρηση που θα γίνει το 2023 και που επιτρέπει πιθανές προσαρμογές όπου αυτό είναι απαραίτητο. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες τις οποίες θα ήθελα να επανέλθω. Κατηγορία 3. Ξέρετε ότι η ορολογία, η διεθνής, δίδει τοπική σημαντική σημασία στην κατηγορία 3 και διεθνή σημασία στις θαλάσσιες οδούς από 4 μέχρι και 5. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το επίπεδο λοιπόν των θαλασσίων αυτών οδών έτσι ώστε να παρέμβουμε με τα περιορισμένα χρήματα που έχουμε στις, στα δίκτυα τα οποία παρουσιάζουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εν πάση περιπτώσει η έκθεση της Επιτροπής σας υπογραμμίζει ότι τα TEN είναι αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Χωρίς τα TEN δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Προσπαθούμε τα τελευταία 20 χρόνια τα TEN αυτά να λειτουργήσουν σωστά και νομίζουμε ότι η σωστή και <clears throat> συγκεκριμένη πρόταση είναι θετική. Ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη και όσους άλλους έχουν συνεισφέρει στην προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτερς. Καλό ήταν που ήσασταν εδώ. Κύριε Κοφεράτη, θέλετε πάλι τον λόγο. Θέλετε να σχολιάσετε αυτά που είπαν οι άλλοι σκιώδεις και η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όπως είπα, επιφυλάσσομαι να συνεργαστώ με τους κοιόδης εισηγητές και να καταλήξουμε στους πιο, ε, θα έλεγα, αποτελεσματικούς συμβιβασμούς. Πάντως να επανέλθω σε λίγα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι ο προληπτικός διάλογος είναι πάρα πολύ θετικός ιδιαίτερα όταν πρόκειται ε, να χρησιμοποιηθούν κάποιες επενδύσεις, κάποια μέσα, τα οποία τροποποιούν την καθημερινότητα αυτών οι οποίοι έχουν ενισχύσει, θα έλεγα, έχουν αλλάξει με σημαντικό τρόπο την, ε, τις συνθήκες στην περιοχή. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε συνεπώς στους κατοίκους μιας περιοχής και μιας κοινότητας κάποια θέματα, κάποια μέτρα. Θα πρέπει να τα συζητάμε μαζί τους και ο διάλογος αυτός ο προληπτικός εφόσον είναι σωστά οργανωμένος δίδει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, δημιουργεί συνενέσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και το λέω και στη συνάδελφο Χάνσλιτ della Shadow del PPE, eh, la collega Ivanova. E io credo esattamente come lei che bisognerà. Νομίζω ότι εδώ στη φάση που διευκρινίζουμε την πλατφόρμα για τα TNT θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους χρήστες βασικά. Αυτό είναι το καθοριστικό. θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα συνολικά εάν έχουμε σωστούς ορισμούς τις σχέσεις ανάμεσα στους χρήστες και τα δίκτυα. Κατανοώ τα προβλήματα τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κατανοώ αυτά που είπε και για τις προθεσμίες, για τα θέματα της διακυβέρνησης και δεν θα πρέπει πράγματι να αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τους επιτρόπους. όπως μας συμβουλεύει και ο κύριος Όλε Σμίτ από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να εξαφανίσουμε θα έλεγα τις προθεσμίες αυτές και τις δεσμεύσεις τις οποίες αντιπροσωπεύουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με πολύ πραγματιστικό τρόπο τις δυνατότητες που έχουμε και να μην αποκλείσουμε μορφές ευελιξίας χωρίς να θέσουμε υποσυζήτηση τα αποτρεπτικά μέτρα τα οποία θα έλεγα αποτελούνται ουσιαστικά από τις προθεσμίες που έχουμε μπροστά μας στους συγκεκριμένους τομείς. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, Τις λεπτομέρειες θα τις ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των επομένων ημερών. Θέλω να, να ευχαριστήσω λοιπόν όσους με βοήθησαν στο πρώτο κομμάτι της προσπάθειας που έγινε, που ήταν ιδιαίτερα απαιτητική θα έλεγα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την καθοδήγησή σας. Η προθεσμία είναι να ψηφίσουμε στις 11 Οκτωβρίου και να γίνει δεκτή στην Επιτροπή Μεταφορών στις 15 Νοεμβρίου. Θα έχουμε προθεσμία την 10, για τους συμβιβαστικές τη 10 Οκτωβρίου. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις, θα μας ενημερώσει ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που ήταν μαζί μας. Καλώς είναι 5 η ώρα και περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Καλωσορίζω τον κύριο Τζουβά. Θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Mm. θα μας μιλήσει για την συμβάσεις παραχωρήσεων. Uh, Υπάρχουν αρκετοί σκιώδεις εισηγητές όπως εγώ, ο Παντζέρη right? και η κυρία Ρούλε είναι επίσης παρούσα. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ο κ. Γκούσταυσον. Υπεύθυνη από πλευρά Επιτροπή είναι η κυρία Τσισκόφσκα. Θα της δώσω το λόγο αφού ακούσουμε τις απόψεις του εισηγητή. Κύριε Ζουβέ, ε, θα σας δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από το Συμβούλιο. Όχι. Κύριε Ζουβά, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε το έργο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συζητήσουμε λοιπόν το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν εδώ και σε πολλές άλλες, ε, σε πολλά άλλα φόρα, γιατί πρόκειται για ένα θέμα δύσκολο και περίπλοκο. Έγιναν δύο συναντήσεις στις 6 και στις 10 Φεβρουαρίου, στις 21 Μαρτίου και έγιναν και κάποια workshops μετά από την πρόταση του Μάλκολμ και τελικά έχουμε προχωρήσει θα έλεγα σε μια ορίμανση του θέματος στα πνεύματα όλων και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το περίπλοκο αυτό θέμα. Μπορέσαμε να προχωρήσουμε λοιπόν με τις δυσκολίες που αντιπροσωπεύει το θέμα και με όλους όσους εξέφρασαν ενδιαφέρον. Πρώτα κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα μας έδειξαν την δυνατότητα να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας και σε σχέση με τις συμβάσεις παραχώρησης για τα έργα υπάρχει ένα νομικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, για τις υπηρεσίες όχι όμως, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και η απλή εφαρμογή της συνθήκης έθετε προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ταυτόχρονα, πολλοί θα συμφωνήσουμε στην ανάγκη μιας μη παρεμβατικής αντιμετώπισης, κάτι το οποίο απαιτεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για να αποφύγουμε διαφορετικές ερμηνείες, αλλά και ένα πλαίσιο το οποίο να μην δημιουργεί επιπλέον περιπλοκές, να μην αυξάνει το κόστος και να μην λειτουργεί εις βάρος του συμφέροντος και των δημοσίων αρχών που εκχωρούν τις ε, συμβάσεις αυτές, αλλά και των οικονομικών εταίρων οι οποίοι έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Το σχέδιο έκθεσης, το οποίο έχω την τιμή να σας υποβάλω, είναι κάτι το οποίο θα έλεγα αλλάζει ε, σε βάθος το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές οι οποίες με ενέπνευσαν. Η πρώτη μας προσπάθεια είναι να διευκρινίσουμε απλοποιώντας την οδηγία. Το κείμενο έγινε πιο ευανάγνωστο και πιο συνεκτικό νομίζω. Βέβαια δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο μου ζητήσατε. Πάντως αυτή ήταν η προσπάθεια την οποία κάναμε. Η δεύτερη βασική αρχή είναι ότι θελήσαμε να επιβεβαιώσουμε τον ειδικό χαρακτήρα που έχουν ε, οι ε, συμβάσεις παραχώρησης σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Δεν είναι μια απλή δημόσια προμήθεια. Και μετά από όλες τις συναντήσεις αυτές που κάναμε, καταλήξαμε στην έννοια α, λεγόμενης ατελούς συμβάσεως. Η ατελή σύμβαση οφείλει να επανεξεταστεί και πολλές φορές οι συμβάσεις παραχώρησης έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μια σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα και που θα ισχύει για 50 χρόνια είναι υποχρεωτικό να αναθεωρείται. Δεν μπορεί να είναι τόσο δίσκαμπτο και σκληρό όσο ε, μια σύμβαση για μια δημόσια προμήθεια. Ε, οι καθηγητές ε, δημοσίου δικαίου μας εξήγησαν ότι το 80% των συμβάσεων ε, των συμβάσεων παραχωρήσεων έδειξαν ότι μέσα σε διετία το 80% των συμβάσεων αναθεωρούνται διότι οι συμβάσεις αυτές εκφύσεως είναι ατελείς και αναθεωρήσιμες. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να υπάρχει πλήρης ελευθερία των δημοσίων αρχών για την επιλογή του νομικού πλαισίου θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε το κείμενο να μην ερμηνευθεί σαν μια επιθυμία ε, ε, ε κρυφής ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών και ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρήσουμε ε, την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία από τη μία και στην ελευθερία από την άλλη ε, των δημοσίων αρχών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραμείνει λοιπόν αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών και δεν θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την έννοια της ατελούς συμβάσεως, λοιπόν. Έχουν καταργηθεί τα ενδιάμεσα στάδια και η διάρκεια της ε, συμβάσεως έχει πλέον διευκρινιστεί και προσπαθούμε τις συμβάσεις αυτές να τις καταστήσουμε πιο ευέλικτες. Τώρα, με την δυνατότητα διατήρησης των κριτηρίων ποιότητας είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ευελιξία και διαφάνεια, εγγύηση φυσικά της διαφάνειας, κατάργηση κάθε περιττής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Θέλουμε γενικότερα να καταστήσουμε τα πράγματα, θα έλεγα, λιγότερο ε, δίσκαμπτα διοικητικά. Θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να μπορούν να επιλέγουν εφόσον το επιθυμούν κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Έχουν υπάρξει κάποιες προσθήκες οι οποίες δεν έχουν υπογραμμιστεί αρκετά. Και γενικά όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν τους κοιόδης εισηγητές. Θέλω να ευχαριστήσω και ε, τους υπεύθυνους για τις νομοδοτήσεις. Έχω τέσσερις ήδη στη διάθεσή μου και περιμένω άλλες δύο. Και νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι δεν θα πρέπει να μακρηγορήσω άλλο. να πω ότι είχαμε πολλές δυνατότητες σε σχέση με το κείμενο αυτό. Κάποιοι πίστευαν ότι θα πρέπει να απορριφθεί το κείμενο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να του δώσουμε κάποιες δυνατότητες, καθιστώντας το πιο ευανάγνωστο, πιο απλό. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, πρέπει οι ρυθμίσεις αυτές να βοηθούν τις ευρωπαϊκές αρχές και φυσικά ε, τους οικονομικούς εταίρους οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Ε, μακρηγόρησα. Πάντως να πω ότι υπάρχει ένα τεχνικό σημαντικότατο θέμα, μείζον θέμα. Διατύπωσα την έκθεσή μου στα γαλλικά, αυτό δεν σας εκπλήσει, και μεταφράστηκε με πάρα πολλά λάθη, τα οποία είναι λάθη ουσίας δυστυχώς. Ε, υπάρχουν παράγραφοι ολόκληροι που έχουν ε, αφαιρεθεί και ταυτόχρονα τα αγγλικά χρησιμοποιούνται σαν βασική γλώσσα. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι ουσιαστικό γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι εργάστηκαν σε ένα κείμενο που δεν είναι το γαλλικό και ε, θα έχουν ένα κείμενο το οποίο ε, δεν περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά. Κατάλαβα λοιπόν ότι το αναθεωρημένο πλέον αγγλικό κείμενο είναι σχεδόν διαθέσιμο, θα το έχουμε στη διάθεσή μας αύριο και θα ήθελα να επιμείνω σε όλους τους συναδέλφους έτσι ώστε τα κείμενα που μεταφράζονται από το αγγλικό κείμενο να αναθεωρηθούν και αυτά, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Λυπάμαι για αυτήν την δυσκολία για την οποία δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Πιστεύω λοιπόν να λυθεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Και τέλος, σε σχέση με το νέο αγγλικό κείμενο, Θα ήθελα να πω ότι το νέο αγγλικό κείμενο δεν έχει διαβαστεί και ελεγχθεί πλήρως από τους ε, νομομαθείς μεταφραστές, αλλά από τα μέλη του γραφείου μου που γνωρίζουν την αγγλική καλύτερα από μένα, αλλά δεν είναι νομομαθείς. Και γι' αυτό λοιπόν η δυσκολία αυτή θα πρέπει να ξεπεραστεί. Το κείμενο είναι από μόνο του ιδιαίτερα περίπλοκο και δεν θα πρέπει να του προσθέτουμε σημεία έλλειψης κατανόησης. Λοιπόν, με την προειδοποίηση αυτή, είδα το κείμενο στα αγγλικά και έχω και ε, κάποιες ερωτήσεις, αλλά η παρουσίασή σας ήταν σαφής, κάνατε μια συγκεκριμένη και πλήρη προσπάθεια. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ζουβά για την ε, δουλειά που έκανε και για την ε, ε, διάθεση και το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε απέναντι στους κοιόδης συζητητές. Θα ήθελα να εκφράσω μια θετική εκτίμηση για την έκθεση αυτή, γιατί αυτή η δουλειά αναδιοργάνωσης και απλοποίησης του κειμένου είναι Περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που τράβηξαν την, το ενδιαφέρον μας ε, ώστε να φτιάξουμε πιο σαφείς ε, ορισμούς και ένα, μια μέθοδο υπολογισμού πιο απλοποιημένη. Μένουν όμως άλλες στοιχείες όπου θα πρέπει περαιτέρω να εμβαθύνουμε. Τα θετικά στοιχεία λοιπόν, καταρχήν η αρχή της ε, διοικητικής αυτονομίας των δημοσίων αρχών και άρα της δυνατότητας των αρχών να αποφασίζουν για τον τρόπο διαχείρισης, για την εκτέλεση εργασιών και την παροχή ε, υπηρεσιών και σύμφωνα με τις αρχές όπου, την αρχή όπου η οδηγία δεν ισχύει σε παιδεία όπου ρυθμίζονται από άλλες τομέακες οδηγίες. Θετική επίσης είναι η διευκρίνηση των ορισμών παραχώρησης για υπηρεσίες εργασίες που τις καθιστά αφέστερες, όπως νομίζω πως είναι καλή και η εργασία συστηματικοποίησης των διαφόρων ορισμών, υποψήφιος, ε, πάροχος ε, κτλ. κτλ. Ε, Επίσης είναι θεμητός και θετικός, θετική μάλλον η αναφορά στις άγνωστες παραμέτρους της αγοράς. Επίσης, η ενσωμάτωση των άρθρων 5 και 7 όσον αφορά την υπολογισμό της αξίας της παραχώρησης με βάση τον κύκλο εργασιών του παραχωρώντος σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν και τέλος θετική προσέγγιση και για τα ε, διατάξεις που σχετίζονται με την παρα... τις παραχωρήσεις in-house, αν και για το θέμα του in-house ίσως θα μπορούσαμε να πούμε κάποια περισσότερα στοιχεία. Να σταθώ μόνο σε κάποια σημεία που θεωρώ πως πρέπει ακόμα να τα δουλέψουμε για να ολοκληρωθεί καλύτερα το κείμενο. Καταρχήν, ε, δεν θεωρούμε σκόπιμη την κατάργηση στην αναφορά στον κύκλο ζωής. Ε, θεωρούμε πως είναι πιο σκόπιμο να προχωρήσουμε σε μια απλοποίηση, ενώ η έννοια θα πρέπει να παραμείνει. Ε, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και θα πρέπει να καταργηθεί και το παράρτημα... Θα, δεν θα πρέπει μάλλον να καταργηθεί το παράρτημα 2. Κάτι που συνδέεται με αυτή την πτυχή είναι ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το κριτήριο της πιο πλανεκτικής οικονομικά προσφοράς, γιατί νομίζω πως πρόκειται για μια, σε ένα σημαντικό ορισμό πάνω στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Περισσότερη δε στένος όσον αφορά τα κριτήρια, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα εργασιακά που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές και εθνικές σχετικές συμβάσεις καθώς και από τις συλλογικέ συμβάσεις. Θα πρέπει όλα αυτά να ξεκινούν με βάση τη διαδικασία την παραγωγική που να είναι βιώσιμη όπως αυτή ορίζεται στην έκθεση Ταραμπέλα και κυρίως αν σκεφτούμε ότι όλα αυτά, αυτές οι παραχωρήσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 35. Υπάρχουν τώρα και συγκεκριμένες παρατηρήσεις τεχνικής φύσης που είναι σημαντικά στοιχεία γιατί επιτρέπουν αντικειμενικά να υποδείξουμε ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ε, θεωρούμε πως είναι αναγκαστική η unblock κύρωση του άρθρου 32 και του άρθρου του σχετικού στο παράρτημα 8 χρειάζεται να διασωθεί τμήμα του άρθρου 32 ενδεχομένω για να εγγυηθούμε τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της κατανόησης και να διευκολυνθεί η μετακίνηση του περιεχομένου στο παράρτημα 7. Σε σχέση με τα άρθρα 35 και 37 θεωρώ ότι η ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων με διάφορους τρόπους θα πρέπει να οριστεί σε αυτό το πλαίσιο ανάμεσα στις ε, ε, ρήτρες εξαίρεσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή, καθώς και η συμμετοχή στην ε, εκμετάλλευση των του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και της παιδικής εργασίας. θα πρέπει επίσης να υπάρχει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την αλυσίδα. Αυτά είναι συνοπτικά τα θετικά στοιχεία που υπογραμμίσαμε, αλλά και κάποια σημεία που πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση, στην καλή δουλειά που έκανε ο εισηγητής κ. Ζουβέν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Κύριε Μάντες, ευχαριστώ και πάλι για λογαριασμό του κυρίου Μπούσολ τώρα. Εάν είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Ζουβά, ότι το αγγλικό κείμενο δεν είναι ορθό, τότε αυτά που θα αναγνώσω ίσως είναι ανοησίες, γιατί βασίζονται στο κείμενο αυτό ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει εγώ θα τα διαβάσω. Let me check, here, um, Mr. Ο κ. Μπούσοικ υποστηρίζει πολλές από τις ιδέες του κ. Ζουβά. Την προσέγγιση για παράδειγμα του εισηγητού που προβλέπει περισσότερη ευκαμψία υπέρ των ε, δημοσίων αρχών και μέσα στα πλαίσια βέβαια των διατάξεων περί διαφάνειας. Ο κ. Μπουσόικ χαίρεται για τις ευκρινήσεις του εισηγητού για την ελευθερία διαχείρισης των, ε, ε, των διοικητικών αρχών, των εθνικών διοικητικών αρχών. Χαίρεται που ο εισηγητής προσπαθεί να διευκρινίσει τους ορισμούς γενικά. για τις παραχωρήσεις και για σημαντικούς επιχειρησιακούς κινδύνους. Ο συνάδελφός μου θεωρεί ότι είναι καλή η εργασία του εισηγητού που διευκρινίζει τι είναι ουσιώδης ε, επιχειρησιακός κίνδυνος, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση όρων όπως operational risk που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στη νομική ορολογία και να προκαλέσει επομένω πολλά προβλήματα. Ένα άλλο θέμα για τον κύκλο ζωής. Εδώ κάνουμε περίπου τις ίδιες παρατηρήσεις όπως ο κύριος Παντζέρη, διότι εδώ έχει διαγραφεί τώρα η οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά. Τώρα για, την, ε, για τον αποκλεισμό ορισμένων δημοσίων φορέων. Χαίρεται ο κ. Μπουσόη για, τα, για την επαναδιατύπωση των άρθρων για τον αποκλεισμό καθώς και για τον αποκλεισμό υπεργολάβων αλλά θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια εξαίρεση in για το άρθρο 15 και για την ανάθεση έργων σε νομικές οντότητες που διεξάγουν όλες τις δραστηριότητε και όχι μόνο το 90%. Ο εισηγητή διατηρεί το άρθρο 2 παράγραφος 15 που ε, έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, περισσότερες συμβάσεις θα αποκλείονται από την ε, από τον ανταγωνισμό, κάτι όμως που έρχεται σε αντίθεση με το στόχο της νομοθεσίας αυτής και για τη διάρκεια θεωρεί ότι η πρόταση του εισηγητού για την διάρκεια των παραχωρήσεων είναι ορθή, είναι σημαντική για να διατηρηθεί η έννοια του κινδύνου στις συμβάσεις που είναι ορισμένου χρόνου. Και επειδή οι συμβάσεις παραχωρήσεων είναι ατελείς, είναι σημαντικό να υπάρξει κάποια ευκαμψία για την τροποποίησή τους. Και γι' αυτό ο Χριστιανό Χριστιαν Μπουσόη χαίρεται για την προσέγγιση του εισηγητού και είναι διατεθειμένος στη βάση αυτή να συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, thank you very much. And um, look forward to... Ωραία. Θα αναμένουμε λοιπόν τη συνέχιση των προσπάθειών. φύγονται από την ιστορία αυτής της αναθεώρησης τρία άρθρα που νομίζω δεν τροποποιούν ιδιαίτερα ε, τις προτάσεις που κάνει ε, ο κύριος Ζουβά. Η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή Ριτά και για την θαυμάσια συνεργασία διότι η συνεργασία αυτή ήταν ανοιχτή και διαφανής και βεβαίως κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα δεν θα εκπλαγεί που θα του πω ότι δεν με έπεισε απολύτως. Θα υποβάλω μια τροπολογία για την απόρριψη συνολικά της προτάσεως της Κομισιόν, διότι θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα δυσχεράνει την ανάθεση ε, συμβάσεων. Θα τις κάνει πιο ακριβές, πιο δαπανηρές δηλαδή, θα αυξήσει το διοικητικό κόστος που κατά μέσον όρο είναι 30.000 σε ολόκληρη την Ευρώπη ευρώ και θα δυσχεράνει και την συμμετοχή διαμεθοριακά που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 1,5%. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου έχω μεγάλες αμφιβολίες διότι έχοντας υπόψη την 40 ετή εμπειρία από την υπόθεση αυτή θα δούμε ότι είναι ένας τομέας όπου είναι νομικά ιδιαίτερα αμφισβητούμενος και δικαστικά δηλαδή γίνονται πάρα πολλές αμφισβητήσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι διατάξεις αυτές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και επομένως σε λιγότερες δικαστικές διαδικασίες. Δεν έχει πολύ νόημα λοιπόν να επιβαρυνθούν, να δυσχερανθούν οι δημόσιες αναθέσεις με μια πρόσθετη οδηγία. Υποθέτω ωστόσο ότι θα υπάρξει ή ίσως υπάρξει κάποια πλειοψηφία υπέρ των ε, συμβάσεων παραχωρήσεων και γι' αυτό είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ σε ρεαλιστική βάση στην βάση των προτάσεων του εισηγητού. Θα κάνω βεβαίως τροπολογίες. Ένα βρίσκω πολύ καλό, ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που μέχρι τώρα πάντοτε έχω επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έλαβε υπόψη επαρκώς τις διατάξεις της συνθήκης Λισαβόνας και τις επιπτώσεις που έχουν στην ανάθεση συμβάσεων παραχωρήσεων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Βρίσκω καλό ότι τονίζει την ελευθερία διαχείρισης του θέματος από τις ε, τοπικές αυτές αρχές, καθώς επίσης προβαίνει και σε ορισμό των συμβάσεων παραχωρήσεων, κάτι που δεν έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκανε τον κόπο επίσης να αναφέρει και το θέμα των ατελών συμβάσεων με τρόπο κατανοητό. Βέβαια, εδώ δεν συμφωνώ με τον Σάντον των Σοσιαλιστών. Δεν νομίζω, ειδικά για τι συμβάσει παραχωρήσεων, να μπούμε σε τόση λεπτομέρεια στι τεχνικέ προδιαγραφέ. Όλοι οι δήμονε μα είπαν ότι οι συμβάσει παραχωρήσεων έχουν κάποιο νόημα όταν πρόκειται για μια light approach. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Οι παραχωρήσει χρειάζονται μια ήπια προσέγγιση. Έχω δε δύο θέματα τώρα όπου αντιμετωπίζω προβλήματα με την πρόταση του εισηγητού και θα σας τα πω. Το πρώτο είναι η ανάθεση κοινωνικών συμβάσεων που το βάζετε στις αιτιολογικές σκέψεις. Όλοι θυμούμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι αν κάνει σχετικέ προτάσεις θα εξαιρέσει ρητά τις συμβάσει αυτέ. Δεν το έπραξε. Εσεί τα έχετε βάλει στα recital, στι αιτιολογικέ σκέψει. Αυτό δεν αρκεί. Διότι εσεί το αιτιολογείτε με, την, με το χαμηλό κόστο. Όμω εδώ πρόκειται και για υπηρεσίε διασώσεω, οι πυροσβεστικέ υπηρεσίε που είναι πολύ μεγάλη αξία και δεν πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Το δεύτερο σημείο που με απασχολεί, και εδώ βεβαίω υπάρχει και άλλη έκθεση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών όπου την έχει κάνει ένας Ολλανδός εισηγητής, ο κύριος Κόλ. Αν συγκρίνει κανείς αυτή την έκθεση με την έκθεση Ζούβα, βλέπει ότι η έκθεση Ζουβά επηρεάζεται ιδιαίτερα από εθνική ε, σκοπιά, γιατί εξαιρεί, για παράδειγμα, τις ηλεκτρικές, τις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή βγάζει τελείως το ηλεκτρικό ρεύμα απ' έξω. Κάτι που ε, ταιριάζει απολύτως στο γαλλικό μοντέλο που δεν έχει, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως απελευθέρωση εκεί. Ο κύριος Κόλ της Επιτροπής Περιφερειών εξαιρεί τις υπηρεσίες παροχής ύδατος και αυτό εντάσσεται στην Ολλανδική νοοτροπία, άλλωστε και στη Γερμανική. Ενώ ο κύριος Ζουβάν θεωρεί ότι δεν μπαίνει το νερό εδώ. Ο κύριος Κόλ το βλέπει διαφορετικά. Γι' αυτό και θα πω ότι νερό, υπηρεσίες διάσωση, πυροσβεστικές και άλλες, πρέπει να συζητηθούν, καθώς επίσης και το θέμα των παραχωρήσεων, των συμβάσεων των παραχωρήσεων για την ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόλε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα σαν σκιώδης της ομάδας μου. Να πω ότι τελικά η στάση την οποία κρατά ο κύριος Ζούβα είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε προσπαθεί να διευκρινίσει, να αναδιοργανώσει και να απλοποιήσει την οδηγία έτσι ώστε να το καταστήσει ένα πραγματικό μέσο αποτελεσματικό. Μην ξεχνάμε ότι τι πρέπει να είναι ε, η νομοθεσία γύρω από τις δημόσιες προμήθειες. Ένα νομικό μέσο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια έτσι ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές χωρίς διακρίσεις, με μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία προς όλους τους συμμετέχοντες και ε, με ξεκαθαρισμένες διαδικασίες. Προς στιγμή λοιπόν το θέμα με τις συμβάσεις παραχώρησης είναι ότι ο ορισμός των παραχωρήσεων, των συμβάσεων παραχωρήσεων ποικίλει, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες είναι κάτι το πάρα πολύ προχωρημένο, σε άλλες χώρες δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, σε κάποιες χώρες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς και όχι σε άλλους. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι η οδηγία αυτή να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις τοπικές ανησυχίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν οι τοπικές αρχές και ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να ε, συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Ο εισηγητής έκανε λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουμε το τι είναι μια σύμβαση παραχώρησης. Νομίζω ότι τον να ασχολείται κανείς με το ότι μια σύμβαση παραχώρησης από τη φύση της είναι μακροπρόθεσμη είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα τύχει τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής, της ισχύω της συγκεκριμένη οδηγίας και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Εδώ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά λοιπόν Ο εισηγητής. Έχει σημασία λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τη φύση των συμβάσεων αυτών. Ο κύριος Παντσέρη πάρα πολύ σωστά είπε ότι οι προτάσεις τις οποίες έχει κάνει ο κύριος Ταραμπέλα σε σχέση με την οργάνωση των συμβάσεων και τα κοινωνικά επίπεδα που πρέπει να γίνονται σεβαστά θα πρέπει να ισχύσουν εκ νέου. Έχει σημασία βέβαια και το είπαν όλοι οι ομιλητές να θεωρήσουμε ότι οι συμβάσεις παραχώρησης είναι ένα εργαλείο ε, για τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πρέπει εμείς να προσθέσουμε ρυθμίσεις οι οποίες ε, καθορίζονται από, τις, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, για τις συμβάσεις εργασίας όπως την απαγόρευση της παιδικής απασχόλησης. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε με αφορμή αυτή τη ρύθμιση ένα μέσο για να ενισχύσουμε αν θέλετε τα εργασιακά ε, υπέρ των εργαζομένων στις διάφορες χώρες. Αυτά θα τα αντιμετωπίσει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, τα διάφορα κράτη-μέλη και όχι η συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό αναλυτικότερα στα πλαίσια της κανονικής διαδικασίας. Πρέπει λοιπόν η πρότασή μας να είναι συμβατή με τα ισχύοντα και σε σχέση με τις υπεργολαβίες που είναι και ένα διαχειριστικό μέσο για τους συμμετέχοντες, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίζουν αυτοί οι οικονομικοί εταίροι. Γιατί αυτό το οποίο μετράει τελικά είναι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Υπάρχει ένα επιπλέον θέμα σχετικά με την ποιότητα, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την επίτευξη των στόχων. Πολλά από τα κριτήρια τα οποία εμπλέκονται στις ε, συμβάσεις παραχώρησης συνδέονται με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Και ο συμβαλόμενος μπορεί να συμπεριλαμβάνει και στόχους ε, σαν παράδειγμα για την επίδοση της υπηρεσίας, για την απόδοση της υπηρεσίας, για τη διαθεσιμότητα στον χρόνο της υπηρεσίας. Κάτι το οποίο ίσως εδώ να μην μπορεί κανείς να το ξεχωρίσει από μια ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά δημόσιες προμήθειες. Αυτό το έχει ε, ρυθμίσει ο κύριος Ζουβά λοιπόν και μπορεί να συμπεριληφθεί. Και εφόσον λοιπόν η εθνική νομοθεσία γίνεται σεβαστή, θα πρέπει ο εργολάβος σε εισαγωγικά να προκρίνει αυτός το είδος και τη μορφή της διαχείρισης ε, την οποία θα επιλέξει για να τρέξει το έργο. Λοιπόν, έχει ήδη συμφωνηθεί με τον κύριο Ζουβά και τους σκιώδης εισηγητές ότι χρειάζεται χρόνος χρειάζονται κάποια εσωτερικά σεμινάρια, χρειάζεται περαιτέρω εξέταση των συμβάσεων παραχώρησης. Το κάναμε αυτό, ήταν απαραίτητο, είναι κάτι το διαφορετικό από μια απλή δημόσια προμήθεια. Και ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει ότι υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην πρότασή της έτσι ώστε η πρόταση αυτή να είναι αποτελεσματική, εύχρηστη και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία επιθυμούμε, επιτρέποντάς μας παράλληλα την χρήση των συμβάσεων παραχώρησης με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Αυτά. Η κυρία Φερχάιεν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ζουβάν για την επικοδομητική συνεργασία για την σύνταξη του σχεδίου εκθέσεως. Είναι σπάνιο πραγματικά να προσφέρει ένας βουλευτής τέτοια συνεργασία που βεβαίως είχε και διαφορές απόψεων, αλλά είναι πολύ σημαντική σε αυτά τα θέματα των συμβάσεων παραχωρήσεων, διότι οι καταστάσεις στις ε, χώρες μέλη είναι πολύ διαφορετικές, καθώς και οι δομές που έχουν δημιουργηθεί διαφορετική μορφή, καθώς επίσης οι επιπτώσεις που έχουν διαφορετικές συμβάσεων έχουν ε, μεγάλες διαφορές. Θα υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Ρούλε και από τη δική μας σκοπιά, διότι όχι επειδή δεν είναι ορθό το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Ζουβά, αλλά διότι η πρόταση της Κομισιόν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Ούτε, επάσης, ούτε επίσης συγγνώμη, η μελέτη επιπτώσεων δεν είναι επαρκής. Η εντατική αναθεώρηση της προτάσεως αυτής από πλευράς του κ. Ζουβά δείχνει και πόσο μεγάλη ανάγκη είχε από επανεπιξεργασία το κείμενο της Κομισιόν. Το περιεχόμενο της προτάσεως αυτής εφόσον υλοποιηθεί θα σημάνει πολύ περισσότερη επιβάρυνση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Χαίρομαι που ο Φιλίπ Ζουβά στην εργασία του που είναι εξαιρετική έχει περιοριστεί στα ουσιώδη, έχει διαγράψει πράγματα τα οποία είναι περιτά, έστω και αν δύο πράγματα μένουν ακόμα να συζητηθούν. Το ζήτημα των διακοινωτικών συνεργασιών και της ανάθεσης in-house Αυτά θα απαιτήσουν και άλλες συζητήσεις στην διάρκεια της επεξεργασίας της εκθέσεως. Και ιδίω για τις αναθέσεις προσφοράς υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι οι συνήθεις διαδικασίες. Υπάρχουν ειδικέ συνθήκες και ιδίω όταν πρόκειται για την παροχή ή προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών ή για θέματα όπως η ίδρυυση, παροχή οπως η ιδρευση ύδατος κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι σε πολλά μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά ειδικά και σε αυτά που ανέφερε η κυρία Ρούιλε, όπως το νερό, το μέσο του νερού. Πολλές χώρες το νερό το θεωρούν σαν κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή τις παροχές, την παροχή ίδρυυσης. Εκεί χρειάζεται μια σε βάθος συζήτηση που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και σε αυτήν θα συμμετάσχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σικόφσκα για να μας δώσει την αρχική αντίδραση της ε, Κομισιόν στην παρουσίαση στην έκθεση του κ. Ζουβέν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή ΕΜΚΟ, και όλοι όσοι συμμετέχουν ε, και αναγνωρίζουμε πόσο ευαίσθητος είναι ε, αυτός ο φάκελος. Είμαστε ήδη ευγνώμονες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά και η συνεργασία ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά για όλα αυτά. Όπως η Κομισιόν έχει πει επανειλημμένος, Στόχος είναι να βρούμε τη λύση για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης. Και γι' αυτό θέλουμε τόσο η δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο να συγκλίνουν και να στοχεύσουν στην εξέβρεση μιας τέτοιας εναλλακτικής λύσης, ώστε να ότι καλωσορίσουμε και γι' αυτό και καλωσορίζουμε αυτή την ε, προσέγγιση. Επίση, αναγνωρίζουμε τι προσπάθειε που έχει καταβάλει ο εισηγητή για να βρει εναλλακτική διατύπωση για κάποιου ε, διατάξει. Ε, είδαμε ότι έχει υπάρξει πολλή προβληματισμό και πολλή δουλειά πίσω από όλα αυτά. <clears throat> Και το εκτιμάμε ιδιαίτερα αυτό. να πούμε επίσης ότι η οδηγία όπως έχει τώρα έχει απλοποιηθεί και βλέπουμε πως υπάρχει εναλλακτικό τρόπος να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει το κείμενο από τη στιγμή που αυτό θα παρα... θα, θα θέτει ορισμένου συγκεκριμένου στόχου, όπω η ισότητα ευκαιριών, η διαφάνεια, η, ανα η ανοιχτή αγορά και η αποτελεσματική χρήση των χρημάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να είναι λειτουργικό αυτό το ε, κείμενο. Κατά τα άλλα, όλες οι άλλες αλλαγές ε, μπορούν και να μας βρουν σύμφωνος. Να τονίσω τώρα κάποια ε, στοιχεία τα οποία θεωρώ σημαντικά πρώτα απ' όλα αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες πτυχέ που ανησυχούν διάφορους ε, ευρωβουλευτές έχουν διευκρινιστεί και καλωσορίζουμε την πιο ξεκάθαρη αναφορά στις ε, ε, αναθέτουσες αρχές ώστε να μπορούν αυτές να καθορίζουν τον τρόπο μάλλον την διαδικασία για την ανάθεση αυτών των των ε, συμβάσεων. Επίσης θεωρούμε ότι ο ορισμός της ε, ε, παραχώρησης προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να πω επίσης πως η Κομισιόν εκτιμά ιδιαίτερα πως το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν έχει αλλάξει. Η οδηγία παραμένει ένα οριζόντιο μέσο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μείνει έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθεί κανένα τομέα από αυτή την οδηγία. Δεν έχει αποδειχθεί και δεν έχει και υπονοείται ότι υπάρχει λόγος να αποκλείσει οποιοδήποτε τομέας από τους κανόνες της ε, ανάθεσης, ε, της ε, σύμβασης παραχωρήσεων μάλλον, της αδειοδότησης ε, και το είδαμε και γιατί δόθηκαν παραδείγματα για τις αεροπορικές μεταφορές και για τις ε, ε, οδικές μεταφορές επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για την δημόσια συνεργασία. Υπάρχει πλήρης αναγνώριση του υπόθεσης του in-house από το δικαστήριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκτιμούμε πως αυτό έχει μείνει το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό για την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, κάποια ακόμα σημαντικά στοιχεία είναι ότι το κείμενο έχει απλοποιηθεί. Όπως είπα, πρόκειται για μια εξέλιξη αλλά νομίζω πως έχει επίσης γίνει κατανοητό πως είναι ένας τομέας που είναι τόσο περίπλοκος που δεν μπορεί να ρυθμίζεται από 6-7 αρθράκια. Απαιτείται από σαφήνιση ορισμένων νοημάτων, ε, ενιών, ε, ε, από σαφήνιση επίσης υποχρεώσεων και καθηκόντων και πιστεύω πως αυτό είναι η σωστή παράμετρος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Να πω επίσης ότι για τη μελλοντική μας ε, συνεργασία πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα σε οποιαδήποτε περαιτέρω απλοποίηση και την εξασφάλιση του περιεχομένου στις διάφορες διατάξεις γιατί δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε, να, να, να αποκαταστήσουμε το status quo, ε, ενώ αυτό προσπαθούμε όντω να διορθώσουμε. Εντάξει, δηλαδή απλοποίηση, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το νόημα ορισμένων διατάξεων. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο είναι Ε, είναι κάτι άλλο σημαντικό είναι ολοκλήρωση των οικονομικών ε, φορέων. Καλωσορίζουμε δηλαδή την ελευθερία των συμβαλωμένων αρχών να καθορίζουν ε, τις διατάξεις όσον αφορά την ανάθεση παραχωρήσεων, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να υποβαθμίζει τις ε, δυνατότητες των οικονομικών φορέων, αλλά θα πρέπει αντίθετα να τονίζει την σταθερότητα και τη σοβαρότητα της διαδικασίας. Κάτι ακόμα που τονίστηκε από διάφορους ομιλητές είναι το θέμα των αλλαγών, των τροποποιήσεων. Είναι σωστό ότι πρέπει να προβλέψουμε ένα βαθμό ευελιξίας όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη γιατί υπάρχουν ε, τρόποι, μάλλον κανόνες για τις τροποποιήσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία καιροσκοπική χειραγώγηση ε, του, της σύμβασης με στόχο το κλείσιμο της αγοράς. Ευχαρίστως να δούμε περαιτέρω δυνατότητα ανοίγματο και απλοποίηση των κανόνων όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι διατάξει αυτές ε, υπάρχουν για να εξασφαλίσουμε δίκαιη πρόσβαση των ε, φορέων ε, των, παρα, παραχωρήσεων στην αγορά. Και ευχαριστώ να σας δώσουμε συμβουλές ή επεξηγήσεις όπου αυτό χρειάζεται. Και σας ευχαριστούμε για αυτό το κείμενο. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πολύ επικοδομητική σας στάση και για την συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε μια πολύ καλή βάση. Όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε αρκετή δουλειά και ε, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ενδεχόμενες βελτιώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Να δώσω το λόγο στον ε, ιδιαίτερα επιμελή Ζουβά ε, να κάνει τις τελικές του παρατηρήσεις και ίσως και να μιλήσουμε και για το χρονοδιάγραμμα πάλι που έχουμε ε, μπροστά μας. Κύριε Ζουβά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τα επικοδημητικά σας σχόλια. Θα ήθελα να σας πω εν γέννη πως φυσικά θεωρώ προφανώς πως το κείμενο βρίσκεται σε συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης και πρέπει να εξακολουθήσουμε να το βελτιώνουμε. Αυτό εννοείται. Καταρχήν να μιλήσω για τον κύριο Παντζέρη. Ο κύριε Παντζέρη, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τα κοινωνικά περιβαλλοντικά κριτήρια από τα οποία εσείς αναπτύξατε. Θα είδατε, θα παρατηρήσατε ότι επέμεινα περισσότερο από ό,τι στο αρχικό κείμενο. Ε, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Και βλέπουμε σαφώς ότι το κείμενο που θέλουμε να ψηφίσουμε είναι πραγματική συμμετοχή για την κρατική αρχή και για την επιχείρηση που θα έχει την παραχώρηση. Δηλαδή, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι αστεία τέτοια κείμενα ε, δεν, πρόκειται, δεν θέλουμε να έχουμε απλέ ε, δηλώσει προθέσεων. Θα πρέπει να υπάρχουν, υπάρχουν πλεονεκτήματα στι αλλαγέ στα κείμενα, αλλά και πάλι να σα πω ότι είμαι ε, διαθέσιμο. Για την αναφορά στον κύκλο ζωή που αναφέρθηκε από τον κύριο Μάντρε, σα ομολογώ ότι δεν έχω κάποια γενικότερη φιλοσοφία, δεν έχω προκαταλήψει. Μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε. Μπορεί και εκεί να υπάρχουν πλεονεκτήματα. Ο κύριο Μάντρε υπογράμμισε την ε, δυσκολία του νοήματος του κινδύνου εκμετάλλευσης. Ίσως εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Έχω σημειώσει 90 με, 80 με 90% μέχρι και 100% βλέπω πως κάποιοι δεν συμφωνούν γιατί Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που επικρατούν ακόμα και μέσα στην ίδια πολιτική ομάδα και ίσως θα πρέπει να πάρουμε κάποιο χρόνο, να το σκεφτούμε καλύτερα για να βρούμε μια λύση που θα μας βρει όλους σύμφωνους. Πρέπει κάποια πράγματα να διευκρινιστούν βεβαίω. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Ναι, και εντάξει, δεν περίμενα να σας πείσω σήμερα, έχουμε ακόμα χρόνο. Δύο πράγματα όμω θέλω να σας πω. Όταν λέτε ότι η παραχώρηση θα κοστίσει περισσότερο, είναι πιο ακριβή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο έτσι αόριστα, γενικά και αόριστα. Και μου εξήγησαν, ας πούμε, το κόστος του νερού σε παραχώρηση. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό στη Γερμανία και στη Γαλλία. Γιατί το νερό είναι πολύ σημαντικό θέμα και ο κόσμος μας λέει το να δώσουμε το νερό στο, σε παραχώρηση, δηλαδή να το βγάλουμε από την εταιρεία υδάτων και το δώσουμε σε κάποια παραχώρηση, είναι, θα κοστίσει περισσότερο. Ήρθαν και κάποιοι οικονομολόγοι που μας παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για μια ολόκληρη σειρά παραχωρήσεων και μας είπαν το εξής στο, στην ερώτηση του αν το νερό σε παραχώρηση είναι πιο ακριβό για τον καταναλωτή από ότι το νερό στην ε, βασική εταιρεία υδάτων, η πρώτη απάντηση ήταν ναι. Όταν δηλαδή η διαχείριση γίνεται σε παραχώρηση, είναι εν γέννη πιο ακριβό από ότι αν γίνεται από κρατική, την κρατική εταιρεία ιδιάτων. Όμως, Ωστόσο, συγκρίνουμε πράγματα που δεν, μπορούν, δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, γιατί η μελέτη διευκρινίζει παραχωρήσεις που έχουν γίνει και δείχνει ότι σε παραχώρηση περνούν βασικά τα δίκτυα διανομής δικτύου που ιστορικά ήταν λιγότερο συντηρημένα. Άρα λοιπόν αυτά που έχουν ε, σημαντικό κόστος εκμετάλλευσης και αν αφαιρέσουμε αυτή τη σημαντική στρέβλωση και αν δηλαδή ε, συγκρίνουμε δίκτυα της ίδιας ποιότητας, οι οικονομολόγοι μας λένε ότι το κόστος είναι βασικά το ίδιο. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Απλώς διάβασα τα όσα λέγαν όλοι αυτοί οι ειδικοί. Προσπαθώ να μάθω και ε, φυσικά δεν... Ε, και, όσον αφορά το... την ελαφριά προσέγγιση, light, Συμφωνώ μαζί σας, το κείμενο λέει άρθρο 26 ότι η δημόσια αρχή γνωστοποιεί την, την, την πρόθεσή της, δηλαδή ε, εκδίδει μια ανακοίνωση περί παραχώρησης, περνά κάποιο χρονικό διάστημα και αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται ε, υποβάλλουν υποψηφιότητε. Τότε λοιπόν η δημόσια αρχή εξετάζει τους υποψηφίους, ισότιμα, μπορεί να διαπραγματευτεί και μετά ανακοινώνει την επιλογή της. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην ελεύθερη βούληση, το... στη διακριτική ευκαιρία της δημόσιας αρχής. Λέμε πως έχουμε κάποιες αρχές. Δημοσίευση της ε, κοινοποίησης αυτής, της ανακοίνωσης αυτής, Έπειτα θα πρέπει να μελετηθούν όλες οι προτάσεις με τον ίδιο τρόπο, με διαφανή τρόπο. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε και μετά επιλέγουμε. Εγώ αυτή την προσέγγιση επέλεξα στο κείμενο. Και είμαι στη διάθεσή σας ώστε να το κάνουμε και ακόμα πιο light. Αλλά να μην φτάσουμε και σε κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει ισότητα των ε, υποψηφίων, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν παραχωρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όπου τα στοιχεία που καλύπτει η παραχώρηση δίνονται σε ιδιώτες χωρίς όμως επαρκή ισότιμη ε, μεταχείριση. Σε αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε. Και αυτό είναι το κύριο μέλημά μου. Αν όμως νομίζετε ότι μπορούμε με διαφορετικό τρόπο να το καταφέρουμε αυτό και, και απλουστεύοντας ακόμη περισσότερο, ευχαρίστω. vos paroles, je partage votre avis avec l'idée que και κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σας πως η παραχώρηση δεν είναι παρά μόνο ένα εργαλείο, δεν είναι στόχος, είναι ένα μέσο που επιλέγουν οι κρατικές αρχές, οι δημόσιες αρχές, κυρίως οι τοπικές, για να διαχειριστούν μια υποχρέωση που πρέπει να κάνουν. Μπορούν να μην επιλέξουν το κάνουν. Αν θέλουν να το κάνουν, θα πρέπει αυτό να, είναι... Να... Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο συμφέρον, είτε οικονομικό, είτε ποιοτικό, Εγώ ίδιο είμαι δήμαρχο ενό δήμου του, περιοχή του Παρισιού. Πρόσφατα έδωσα μια σύμβαση παραχώρησης για ένα πάρκινγκ γιατί ακριβώ οι δημοτικέ αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν και να διαχειριστούν την εμπορική πτυχή ενός τέτοιου χώρου δεδομένων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ήταν επιλογή διαχείρισης. Κυρία Βερχάγγεν. Σα Σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε την... Ε, το κείμενό μου και εγώ είμαι έτοιμος να προχωρήσω. Αχ, πρέπει να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Θα ήθελα να μπορέσουμε να σαφώς να πούμε πως αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια στη συζήτηση ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους υποψηφίους παραχώρησης. Στόχος είναι να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και νομίζω πως το έχω καταφέρει εδώ και κάποιους μήνες. Θα μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν μια μέση οδό. Είμαι αισιόδοξο. Από ό,τι ε, παρατήρησε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντικατά τη εξέλιξη του κειμένου προ αυτήν την κατεύθυνση και χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης παρατήρησα πως έχετε περιγράψει κάποια στοιχεία που η Κομισιόν, δεν, μάλλον κάποια όρια που δεν θέλετε να ξεπεραστούν από πλευράς Κομισιόν. Θα εμβαθύνουμε σε αυτό. Και νομίζω πως, Πρόεδρε, έχουμε κάνει μακρά πορεία. Έχω την εντύπωση πως κάποιες φορές τα πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά αλλά τους τελευταίους μήνες είδα ότι τα, ε, οι ευρωβουλευτές ε, έδειξαν καλή θέληση ώστε να προχωρήσει το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία από την υποδοχή που έλαβε, που έτυχε η έκθεσή σας σήμερα το απόγευμα. Όλοι στον τομέα, αυτό και στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, δουλεύουν επικοδομητικά έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι πόσο σημασία έχουν. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το κείμενό σας πλέον είναι διαθέσιμο. Θα υπάρξουν κάποιες γλωσσικές ρυθμίσεις στο αγγλικό κείμενο. Πράγματι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα τελικό κείμενο και ευχαριστώ τις υπηρεσίες μας που μας βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή λόγω των αλλαγών που προτείνεται, τις παρακολουθούμε ακριβώς σε ένα τελικό κείμενο. Λοιπόν, προθεσμία 3 Οκτωβρίου 5 το απόγευμα, αυτό μας δίνει ένα μήνα περίπου, χρόνο αν θέλετε, Περίσκεψη 6 Νοεμβρίου, και οι συμβιβαστικές τροπολογίες 28 ή 29 Νοεμβρίου με τελικό στόχο υιοθέτηση 18 Δεκεμβρίου. Περιμένουμε και τις νομοδοτήσεις από άλλες επιτροπές. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον ε, Ιώνας ε, για την προσπάθεια την οποία έκανε. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30. 18, 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και θα συνεχίσουμε εκεί τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει για τις δημόσιες προμήθειες.